να Ε, έχω τη χαρά να καλωσορίζω αντιπροσωπεία της Όιλι ε, που είναι η βολή του Ισπεκιστάν. Έχουμε αντιπροσωπεία ε, στο θεωρείο. Ε, Ζαγρανίτσο, granicą inwestycji τουριστικής, turystyki panem Κουρμανόβεμ Kurmanowem na ο κύριος Αλισερ Κουρμάνοφ είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας αυτής. Με χαρά υποδεχόμαστε την ουσβεγγική αντιπροσωπεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, έχουν έρθει για την 13η συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και με χαρά θα συνεργαστούμε και προσβλέπω σε αυτή τη συνεργασία. Ο κύριος Μπέκερ τώρα για δύο λεπτά παρακαλώ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με